έχω να σας κάνω την ε, λυπηρή ε, ανακοίνωση ότι ο Κίνιος Πέισλι την προηγούμενη Παρασκευή πέθανε σε ηλικία 88 ε, ετών. Ήταν επί μακράων βουλευτής εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο τέλος της θητείας του εδώ πέρα διατέλεσε και υπουργό στην Ιρλανδία. Θα ήθελα κυρίες και κύριοι να σας ενημερώσω ότι πολλοί συνάδελφοι μου επέστησαν την προσοχή το εξής Σήμερα λαμβάνουμε, τώρα δηλαδή που σας μιλάω, λαμβάνουμε νέες δραματικές ειδήσει για ναυάγια, δραματικά ναυάγια. 500 οι ε, θάνατοι εικάζονται στην Μεσόγειο. 36 ενδεχομένως να σωθούν, αλλά ε, περίπου 200 είναι τα άτομα που έχουν χάσει τη ζωή τη, ε, Έξω από τι ακτέ τη μάλτα λοιπόν έχασαν τη ζωή του πάνω από 500 άτομα. Νομίζω ότι έχουμε ηθικό χρέο να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα κυρίε και κύριοι για να προλάβουμε στο μέλλον περαιτέρω τέτοιε ανθρωπιστικέ καταστροφέ τι οποίε δεν μπορούμε πραγματικά να επιτρέψουμε. Κυρίε και κύριοι, την προηγούμενη εβδομάδα σα ανακοίνωσα και θα ήθελα εδώ να το επαναλάβω ότι αύριο, λίγο πριν την ψηφοφορία, εδώ θα γίνει μία μαγνητοσκόπηση, α, συγγνώμη, όχι αύριο, την Τετάρτη, πριν την ψηφοφορία, λοιπόν, 360 μοιρών. Όλα, λοιπόν, τα μέλη θα καταγραφούν με μια τέτοια κάμερα περιστροφική, ξέρετε, λοιπόν.